Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Άρχεται η συνεδρίαση, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Σίμψον. I hope that most members will be able to... Ελπίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα μπορέσουν να με βλέπουν, παρά το ότι μπροστά τους αυτό το βουνό από χαρτιά, κοντά μου λανοξύστης είναι, για τα χαρτιά της συνεδρίασης, Κάνουμε εκείνη τη συνεδρίαση ω ε, πιο νωρί έγινε από το, το Connecting Europe και τώρα ξεκινάμε τη δική μα συνεδρίαση και ξεκινάμε με την έγκριση των πρακτικών. Last Transport Committee meeting, which was on the 8th, 9th of October. Ε, και λέμε τώρα για συνεδρίαση 8 και 9 Οκτωβρίου, αν δεν έχετε κάποια ένσταση για τα πρακτικά, εγκρίνονται. Και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η ανακοίνωση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με την ΕΜΣΑ ή τον ΕΜΣΑ, Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. 25 Οκτωβρίου ε, και λέει ότι αυτή η θέση του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα μας για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, λεφτή απόφαση κατόπιν της ανακοινώση αυτής και θα πρέπει να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η θέση του Συμβουλίου ε, αποκρισταλώθηκε στις 25 Δεκάτου και έχουμε το σχέδιο της σύστασης του κ. Φαγκενστάιν το οποίο θα το συζητήσουμε για την πρώτη ανάγνωση αύριο το απόγευμα. Και επίση σας υπενθυμίζω ότι το κείμενο το οποίο έκανε το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει τη συμφωνία μεταξύ εισηγητού και οδών εισηγητών και του Συμβουλίου, όπω εγκρίθηκε από την Επιτροπή μα στι 24 Τετάρτου ενεστώτο έτου. Και τέλο θα πρέπει να σα πω ότι η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι η 5η 11 στι 12 το μεσημέρι, τόσο ώστε να γίνει η ψήφιση στην Επιτροπή μα στι 27 Ενδεκάτου και να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αυτά για να ξέρετε τι ισχύει για τη θέση του Συμβουλίου. Το επόμενο θέμα τώρα, σας υπενθυμίζω συνάδελφοι, είναι ότι έχουμε παντού αυτή τη βδομάδα τηλεκάμερες. Έχουμε και μετάδοση ζωντανή από το ίντερνετ, οπότε αυτό να το έχετε υπόψη, ότι εκτός από την ιντερνετική μετάδοση έχουμε και την τηλεόραση του Κοινοβουλίου. Εν δράση. Τώρα το επόμενο μας θέμα είναι. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο το απόγευμα θα γίνει η ψηφοφορία. Βέβαια έχουμε ψηφοφορίες και αύριο το πρωί. Άρα. Να έχετε λοιπόν αύριο όλη μέρα τις κάρτες σας, τις κάρτες σας και θα ισχύσουν αυστηρά όλες οι ίδιες διατάξεις και παρακαλώ να έχετε τις κάρτες κάρτες και παρακαλώ οι συνεργάτες των βουλευτών να βοηθήσουν, να εξασφαλίσουν το να έχετε όλοι οι της τις κάρτες σας. Πάμε λοιπόν ευθύ αμέσω στα θέματα 5 και 6 που είναι το θέμα της δέσμης μέτρων για τα αεροδρόμια και τα σχετικά ε, με, τις, με την εκμετάλλευση και έχουμε τον κύριο ή τον κύριο Ζασάντα και οι άλλοι συνάδελφοι θα, θα μας μιλήσουν που έχουν αναλάβει. Ο πρώτος ο κύριος Ζασάντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κύριος Ζασάντα, έχω πω τα εξή. Έχουμε πάνω από 500 τροπολογίες, για τις οποίες ευχαριστώ άπαντες. Ξέρω ότι έχετε καταβάλει σχετικώ πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επεξεργαστείτε τι τροπολογίε αυτέ και αυτές οι 500 συν και πλέον τροπολογίε με οδήγησαν ει 8 ε συμβαστικέ διατάξεις τις οποίες και έχω υποβάλει. Εις τους συναδέλφους που είναι σκιώδεις ηγητές. αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διεκπαιρέωσή μας και έτσι τελικά ελπίζω να τα βρούμε. Πρόκειται για οκτώ σημαντικά σημεία τα οποία μας εδίχασαν στην αρχή αυτής της διαδρομής εδώ τις βασικές πολιτικές περιοχές του Κοινοβουλίου. Φαίνονταν αδύνατον, αλλά μετά από μια σειρά συναντήσεων απεκόπησε την εντύπωση ότι στα 7 από τα 8 αυτά σημεία έχουμε έναν πραγματικό αυθεντικό συμβιβασμό. Επιτρέψτε μου επομένω να αναφερθώ σε αυτά τα σημεία και στο τέλος θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα πιο μεγάλα σημεία. Πρώτα πρώτα ξεκινούμε. Συμβαστική Β αφορά το πώς οι υπηρεσίες εδάφους θα διαχωριστούν από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, τις κυρίες υπηρεσίες του αεροδρομίου. Έχουμε τα εξή πρώτα-πρώτα. Έχουμε την πλήρη 100% ε, και διανόμου ε, διάκριση και διαχωρισμό, τη λειτουργική, του λειτουργικό του με διαχωρισμό, λειτουργικό. Επίσης, από την δημιουργία έχουμε και τον τελικό ε, διαχωρισμό. Αυτά με αυτόν τον συμβασμό. Άρα πρόκειται κατ' ουσίαν για έναν διαχωρισμό που αφορά την διαχείριση αυτών των λειτουργιών. Από μια μεριά λοιπόν θα καταρτήσει τι συμβάσει, ο ένα διαχειριστή, ένα εκπρόσωπο στο αεροδρομίο και θα υπάρχει άλλο που θα καταρτήσει συμβάσει που θα αφορούν τι υπηρεσίε εδάφου. Επίσης εδώ καλύπτονται και οι υπηρεσίε που έρχονται από κάποιε εταιρείε από πόρτα σε πόρτα όπως λέμε. Γιατί αυτέ οι εταιρείε δεν καλύπτονται από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη γνώμη μου, καταφέραμε να άρουμε αυτό το κενό νόμου. Τώρα, συμβαστική δέλτα που αφορά το ότι πρέπει να υπάρχει έγκριση για κάθε περιβαλλοντία. Η συμβαστική έψιλον ε για την έγκριση που αφορά τις εταιρείε υπηρεσιών εδάφου. Που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα αεροδρόμια της Ένωσης. Θέλαμε να παρέχεται αυτή η έγκριση άπαξ και κατόπιν η εταιρεία αυτή να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το οποίο θα ήταν προστιθέμενη αξία. Όμως η πρόταση της Επιτροπής ήταν μάλλον περίπλοκη. Στη συμμετοχή μας διάταξη απλουστεύσαμε τα πράγματα. Και έτσι δεν έχουμε αυτή την περίπλοκη διαδικασία της έγκρισης που ουσιαστικά εμπόδιζε τις εταιρείες από το να παρέχουν πλήρως τις υπηρεσίες τους. Έχουμε τέσσερα μέρου σημεία, τα οποία θα τα εξετάζουμε σε επίπεδο κάθε κράτου μέλου. Πρώτα από τα ασφάλεια, δεύτερον προστασία, ασφάλεια, ή τέλο ασφαλιστικέ υπηρεσίε, ή ασφάλιση. Και οι δεξιότητε, τα προσόντα θα πρέπει να έχουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτέ τι υπηρεσίε. Συντονισμό τώρα των υπηρεσιών εδάφου αυτό αφορά το, τη συμβαστική H ή Ήτα. Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα. Κατόπιν έχουμε την Θ ή G όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο ποιότητος. Εδώ είπαμε ότι έχουμε πραγματικά μια προσθεμένη αξία την οποία οδηγεί η δική μας ε, διάταξη. Αυτό το οποίο θέλουμε εδώ είναι να υπάρχει ποιότητα σε αυτές τις υπηρεσίες, γιατί όταν μιλούμε για απορρίθμιση Πολλέ φορέ αυτό το οποίο γίνεται είναι να έχουμε επιδείνωση του επίπεδου και της ποιότητας, αν εμεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ε, καλύτερη δυνατή ποιότητα. Και επομένω αυτό το, το, το ελάχιστο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, αυτό θα πρέπει να τάσεται από το ίδιο το αεροδρόμιο. Γιατί το αεροδρόμιο ξέρει καλύτερα το τι μπορεί μέσα στη λειτουργία του να υλοποιηθεί. Βεβαίω, ο έλεγχος θα ασκείται από μια ανεξάρτητη αρχή του κράτους μέλους. Εκείνοι θα υποπτεύουν την όλη διαδικασία. Και τέλος, το πιο επιμεχό σημείο είναι η συμβαστική α. είναι σχετική με την απορρίθμιση. Αυτό το οποίο θα με εδώ είναι να υπάρχει πιο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών που παρέχουν τις υπηρεσίες εδάφους. Δεν πρόκειται περί ανταγωνισμού, εάν έχουμε επιλογή κάποιου συγκεκριμένου υποψηφίου και κάποιε εταιρείε κατά το διαγωνισμό που γίνεται και κατόπιν και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Και αυτό το οποίο σας προνέφερα ισχύει κατά μείζωνα λόγο για τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μας πρόταση είναι συμβαστικού χαρακτήρα και συνενώσαμε εδώ τη, τη, σύμφωνη γνώμη των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων και γι' αυτό ελπίζουμε ότι και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε μέχρι αύριο θα έρθουν να συμφωνήσουν. Αυξήσαμε, ανεβάσαμε το σχετικό κατόφλιο. Από τα 5 στα 10 εκατομμύρια. Δύο θα είναι οι σχετικές εταιρείε. Είχα στην αρχή και μετά πήγαμε στις τρεις για τα μεγαλύτερα 7 αεροδρόμια της Ένωσης. Εκεί που είχαμε την πραγματική απελευθέρωση και απορρίθμιση ε, στις υπηρεσίες αυτές και μιλούμε τώρα για 35 εκατομμύρια πλατών ετησίως και έτσι έγινε αυτό το άνοιγμα και είπαμε ότι από τις τρεις μπορεί να μπει και μια τέταρτη σε αυτά τα αεροδρόμια, μια τέταρτη εταιρεία παροχή υπηρεσιών έδαφος. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για το όλο τοπίο που αφορά το ελεύθερο μα Σημαίνει ότι ένα κράτο μέλο μπορεί να έχει ένα ολόκληρο πλέγμα κανόνων και κανονισμών και μπορεί να έχει σε πέντε χρόνια τρεις εταιρείε και κατόπιν να έχει τέσσερις μετά από πέντε χρόνια. Επομένως, αυτό τι είναι, είναι άκρατη φιλευθεροποίηση. Ερωτώ. Από την Ελμυριά, στο Τόκιο, έχουμε δέκα εταιρείε παροχής υπηρεσιών εδάφους. Τρεις είναι ανεξάρτητες από αυτές και δεν προβλέπονται διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες να μπορεί μια αεροπορική εταιρεία να συνάψει μια σύμβαση με κάποια συγκεκριμένη εταιρεία ε, παροχής πλούσιων είναι Όμως εδώ δεν είμαστε Ιαπωνέζοι. Εδώ επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο εμεί μπορούμε να σκαρφιστούμε και να κλείσουμε συμβασμό γιατί εδώ πρόκειται περί συμβασμού. Και έτσι κυρίως θέσεις προσοχή μας στα μεγάλα αεροδρόμια θα είναι μια διαδρομή που θα κρατήσει κάποια χρόνια και θα εξασφαλίσουμε θέσεις απασχόλησης. Η Επιτροπή Απασχόλησης ολοκλήρωσε το δικό της κομμάτι προ ημών και πρότεινε κάποιες λύσεις όσον αφορά τους εργαζόμενους αυτές τις εταιρείες. Πρότεινε κάποιες λύσεις που πουθενά δεν ισχύουν στην Ευρώπη. Και αυτό να το θυμόμαστε. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα τέτοιο άνοιγμα, θα πρέπει να θυμόμαστε τι έχει προταθεί και αυτές τις λύσεις που θα είναι από το τμήμα του εγγράφου, του νομοθετήματος. Γι' αυτό και ε, εκπλήσουμε από κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να απορρίψουν όλο το έγγραφο. Όμως, αν αναπαιθεί το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα έχουμε πρόβλημα και θα ανατραπούν όλα όσα μέχρι τώρα έχει προβλέψει και η Επιτροπή Απασχόλησης. Όλα αυτά τα προστατευτικά μέτρα θα μπουν στο χρονοτούλοπο. Μέσα όλα αυτά τα εξετάζουν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε αυτό το έγγραφο και θα πρέπει τελικά να δούμε πώς θα ξεχάσουμε λένε κάποιες από τι λύσει, γιατί ορισμένοι δεν θέλουν να έχουν αυτή τη λύση σε ένα αεροδρόμιο, Περνάνε 10 εκατομμύρια επιβάτε και έχουμε ε, να έχουμε υγιείς του ανταγωνισμού και αυτοί που θέλουν να λειτουργήσουν το έγγραφο δεν θέλουν. Ε, τέλος πάντων, σας ευχαριστώ και πάλι. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Ίσως είναι οριακές οι πλειοψηφίες αύριο στην ε, ψηφορία. Καλά, θα επεξεργαστούμε και άλλο το έγγραφο, αλλά να το αναπέμψουμε το, το έγγραφο αυτό από την πρώτη ανάγνωση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαίνει ότι θα πάει χαμένη η δουλειά και η δική μας και των άλλων επιτροπών. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Πρώτα θα ασχοληθώ με το θέμα των υπηρεσιών εδάφους και μετά στο θόρυβο. Ο κύριος Μαν της Επιτροπής Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Απασχόληση το Σεπτέμβριο ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξέταση τη έκθεση ακριβώ επειδή διακρίναμε το πρόβλημα αυτό και είχαμε ζητήσει το εξή. Ε, σε όλε τι ε, σκέψει ε, περί απόρριψη τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά το αποτέλεσμα θα ήταν να παραμείνουμε άφωνοι, να μην έχουμε γνώμη και να παραπευθύνει το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρότεινα στους συναδέλφους στην Επιτροπή να ε, φροντίσουν σε κάθε περίπτωση να συζητήσουν τις θέσεις τους για να καταφέρουμε να βρούμε την ε, πλειοψηφία. 36 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Εντάξει, τι να κάνουμε, Μπορεί να μην άρεσε σε όλους αυτή η έκθεση, αλλά δεν αρέσουν όλες οι εκθέσεις σε όλους. Τι να κάνουμε. Αλλά είναι σημαντικό το ότι υπάρχει συμβιβασμός από πλευράς ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Για θέματα εκπαίδευσης θέλαμε σίγουρα να κατοχυρώνουμε τα θέματα αυτά. Και όχι σε μια δύο μέρες όπως ε, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν έχει να κάνει με αρμοδιότητες και σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει ε, του αεροπιβάτη. Αυτό λοιπόν το πετύχαμε. Δεύτερο που πετύχαμε, αν υπάρχει ε, εξαγορά, να παραμείνουν τα δικαιώματα τα οποία έχουν ήδη κατοχυρωθεί. Όπως για παράδειγμα μισθή, όπως ε, συμβάσεις εργασίας και αυτό λοιπόν καταφέραμε να το κατοχυρώσουμε σε κάποια κεφάλαια και υποκεφάλαια για τους ε, αρμόδιους και τους συναρμόδιους. Αλλά σε τελική ανάλωση θα πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε στο Κοινοβούλιο. Ένα ε, άλλο τομέα είναι το τομέα της κοινωνικής ασφάλειας. Ε, είπατε ότι θέλουμε να, το, να την ποιότητα αυτή. Ναι, σύμφωνοι δεν είναι ότι δεν θέλουμε την απελευθέρωση. Κανείς δεν, θέλουμε δεν θέλει να δημορφωθεί ένα μονοπόλιο. Αλλά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και το είχαμε πετύχει στο παρελθόν είναι ότι οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας το οποίο να τηρείται για να μην ε, επιλεχθεί το κριτήριο του ποιος είναι πιο φθηνός. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κοινωνική προστασία Νομίζω ότι πρόκειται ένα από τα πιο βασικά στοιχεία, τα ελάχιστα πρότυπα, οι ελάχιστε προδιαγραφέ. Αυτοί είναι λοιπόν κάποιοι τομεί ε, του οποίου εντοπίσαμε από την Επιτροπή Απασχόληση. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, γιατί νομίζουμε ότι η μεγαλύτερη απόρριψη θα είναι να επιτρέψουμε και άλλους παρόχους χωρίς να ξέρουμε το επίπεδο ποιότητας που θα προσφέρουν και μάλιστα με όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ε, αεροδρομίων. Θα πρέπει να εντοπίζουμε και να λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορές των αερολιμένων και των κρατών μελών. Αυτό μας απασχόλησε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτά λοιπόν, εν μεγάλη συντομία, αυτά που συζητήσαμε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Και φυσικά είμαστε ανοιχτοί προς κάθε συμβιβασμό, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τα πάντα. Και αυτό το κατέδειξε και η διαδήλωση. 2.500 εργαζόμενοι σε αεροδρόμια των ε, αεροδρομίων από όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σαφές μήνυμα, γιατί εμείς οι εκπρόσωποι του λαού θα πρέπει να δώσουμε σαφείς απαντήσεις. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Αρκαντράουι από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώδη εισηγητή Φλέκενστάιν Δυστυχώ αναγκάστηκε να φύγει και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για την προσπάθεια και το έργο του, αλλά θα πρέπει να είμαι και ειλικρινής παράλληλα και να πω ότι ως ομάδα εμείς θα ταχθούμε υπέρ της απόρριψης της πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποτέ δεν ήμασταν ενθουσιώδεις με την πρόταση σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών εδάφους, ιδιαίτερα μετά το 1996 για το άνοιγμα των αγορών και τις συνέπειες των κοινωνικών, ε, στο κοινωνικό τομέα. Αλλά θέλαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο και με τους συναδέλφους και με τους συναδέλφου ε, συναδέλφους από την Επιτροπή την Αρμόδια και θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε κάποια σημεία έχουν γίνει κάποιες μικρές βελτιώσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε όλες τις συμβαστικές ε, τροπολογίες εκτός από την συμβαστική α, που θεωρούμε ότι δεν είναι συμβαστική σε τελική ανάλυση, καθότι δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε. Αυτή η πρόταση πηγαίνει ακόμα πιο πέρα και από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θεωρούμε ότι συνολικά η πρόταση είναι και μη ισορροπημένη και μη κατάλληλη και ανεπαρκή. Θεωρούμε ότι είναι χαμένη ευκαιρία σε ό,τι αφορά κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδο. Δεν επιλύονται σε ό,τι αφορά μεταφορά προσωπικού, ελάχιστους μισθούς, ανακράτος μέλος, που θα μπορούσαμε να τα ορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν δεν πέρασαν. Και για αυτούς τους λόγους λοιπόν όλους θα ταχθούμε υπέρ της απόρριψης της πρότασης. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δεν περάσει η απόρριψη του κειμένου, φυσικά θα υποστηρίξουμε τους συμβιβασμούς που μας βρίσκουν σύμφωνος. Και θα συνεχίσουμε το διάλογο και στην Επιτροπή Μεταφορών, αλλά και στην ε, Ολομέλεια, σε περίπτωση που τελικά ο εισηγητής καταφέρει να πείσει τους συναδέλφους. Φυσικά, στην περίπτωση αυτή θα συμμετάσχουμε στην συζήτηση για να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα στην Ολομέλεια, αλλά όπως έχει το κείμενο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι υποθερίζουμε το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κλέντς για την Άλντε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα ως κοιόδη εισηγητή να πω δύο λόγια. Καταρχά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο εισηγητή ο οποίος κατέβαλε προσπάθεια να συνενώσει Πολλέ και διαφορετικέ απόψει. Αυτό καταδεικνύεται και από τις τροπολογίες, προκειμένου να εξεύρει συμβιβασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την όλη πρόθεση δεν αποσκοπεί σε μια απελευθέρωση ως αυτό σκοπό, αλλά για να βελτιώσει τις υπηρεσίες ε, εδάφους. Εγώ τι να σας πω, αμφιβάλλω κατά πόσον η ποιότητα αυτή εξαρτάται από τον αριθμό των παρόχων. Κοιτώντα ε, τις προσωπικές μου εμπειρίες στο Λονδίνο, στην Ζηρίχη, στο Άμστερνταμ και ούτω καθεξής, τι διαπιστώνω ότι όπου υπάρχει πλήρης απελευθέρωση με 9-10 ε, παρόχους, όπου υπάρχουν 9-10 παρόχοι, δεν είναι καλύτερες και πιο υψηλής ποιότητας οι υπηρεσίες. Άρα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτού κάνει την πρόταση δεν δοκίμασε, δεν ήθελε να δει, δεν εξέτασε κατά πόσον η αύξηση των παρόχων συνεπάγεται και αύξηση της ποιότητα Και συγκεκριμένε προτάσεις. Κοιτάξτε, συμφωνώ με τον προηγούμενο μελητή Σπανίως, σπανίως συμφωνώ σε τόσο πολλά σημεία με εκπρόσωπο των σοσιαλδημοκρατών. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συμφωνώ. Πολλές συμβαστικές προτάσεις έχουν ουσιαστικά διαφορές μόνο στην απόχρωση. Δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Σε ό,τι αφορά την έγκριση των παρόχων. τέσσερα κριτήρια αναφέρονται. Εγώ θα ήθελα να παραμένει και η χρηματοοικονομική ισχύς ως κριτήριο. Δεν θεωρώ ότι σωστά διαγράφει αυτό το κριτήριο του οικονομικού παράγοντα των παρόχων σε ό,τι αφορά το συντονισμό των ε, ελάχιστων προτύπων. Φυσικά και χρειάζονται ελάχιστα πρότυπα, αλλά δεν ξέρω τώρα αν χρειάζονται τόσο εντελεχείς ε, λίστες ε, προτύπων. Αυτό εξαρτάται και από το αεροδρόμιο, για παράδειγμα μπορούμε να ορίσουμε ως ελάχιστο, ελάχιστη πρωτογραφή 30 λεπτά για τον χρόνο μεταβίβασης, μεταφόρτωσης. Αλλά υπάρχουν και διαφορές. Αλλά κοιτάξτε, το βασικό μου πρόβλημα, η βασική μου δυσκολία, συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει όλα αυτά να διαχωριστούν από πλευρά οργανωτική και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα οικονομικό επόπτη, ο οποίο στο τέλη του έτου θα ελέγχει ότι δεν έλαβε χώρα κάποια εγκάρσια επιδότηση. Αυτό είναι σημαντικό και σωστό, αλλά και εμένα με προβληματίζει η συμβιβαστική α. Δεν θεωρώ ότι είναι συμβιβαστική υπέρ της απελευθέρωσης. Εδώ θεωρώ ότι ο συνάδελφος ε, εισηγητής έμεινε στα αρχικά πλαίσια της πρότασης. Εγώ είχα υποβάλει μία συμβιβαστική πρόταση, δεν την έλαβε υπόψη και δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με τη συμβαστική Α εν τέλει. Ευχαριστώ κύριε. Λίχτεμπεργκερ για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, ο οποίος προσπάθησε να εξέβρει συμβιβασμούς, ωστόσο θα πρέπει να ομολογήσω ότι σε ορισμένους τομείς και από δική του ε, πλευρά δεν είχε άλλε δυνατότητε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό σε ό,τι αφορά τι προτάσει τη Επιτροπή Απασχόληση επί του περιεχομένου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσε, αλλά πολύ απλά δεν είναι δεσμευτικέ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πρόκειται για μια γενική διατύπωση, την οποία μπορεί κανεί να τηρήσει, μπορεί και να μην την τηρήσει. Και στην τελική ανάλυση τα πράγματα παραμένουν ως είχαν. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή είναι η δυσκολία. Αν καταφέρναμε ε, να καταστήσουμε τις προδιαγραφές αυτές δεσμευτικές και να μπουν και στην εθνική νομοθεσία, για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένες και τις οδηγίες για τους διαγωνισμούς και τέτοιων άλλων λεπτομεριών. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Κλίνσε, με προβληματίζει το εξής. Δεν πιστεύω ότι είναι και αυτόματο το ότι αν ε, αντικατασταθεί το εθνικό μονοπόλιο με ένα ευρωπαϊκό ολιγοπόλιο θα βελτιωθεί η ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις υπηρεσίες ε, για τις αποσκευές. Ε, χάνονται βαλίτσες και στη Βιέννη και στο Λονδίνο και στην Ιταλία. Άρα, τι να σας πω, τα πράγματα παντού ίδια είναι. Δεν είναι αυτόματη αυτή η αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή ότι με πιο πολλούς παρόχους θα έχουμε και πιο υψηλή ποιότητα. Και θα ήταν ε, πραγματικά ίσως έξυπνο, αν θέλαμε πραγματικά τον επιβάτη να βοηθήσουμε, να κάναμε μία ανάλυση πρώτα ποιοι είναι οι ουσιώδεις παράγοντες που θα πρέπει να αλλάξουν. Κοιτάξτε, επειδή οι κανόνες αυτοί δεν είναι δεσμευτικοί και επειδή ο τέταρτος πάροχος ε, στην συμβιβαστική α μπαίνει από την πίσω πόρτα ουσιαστικά πάλι, αποφασίσαμε να απορρίψουμε την πρόταση θεωρούμε ότι η μοναδική λύση είναι να επαναπεμφθεί αυτή η πρόταση. Αν είχαμε, αν είχαμε καταφέρει που δεν μπορούσαμε γιατί δεν είχαμε τις αρμοδιότητες, αν είχαμε καταφέρει να καταστήσουμε ε, δεσμευτικές τις κοινωνικές τις θα ψηφίζαμε διαφορετικά. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Συστάσεις τώρα. Τι να πούμε, τις συστάσεις δεν ε, πετυχαίνουμε τίποτα. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για στην τελική ανάλυση ο ανταγωνισμός επιβαρύνει και τους ε, επιβάτες αλλά και τους εργαζόμενους. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έκανε τα πάντα, ό,τι μπορούσε έκανε για να μας ε, φέρει σε συμφωνία. Αλλά Ο Πυρήνα έγκυται στην Φραγκφούρτη. Δεν το ανέφερε κανεί. να το αναφέρω εγώ. Οι Γερμανοί συνάδελφοι θέλουν να σπάσουν το μονοπόλιο που επικρατεί στην ε, Φραγκφούρτη. Όλοι στη Γερμανία λοιπόν αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό και γι' αυτό και κάνουμε τη σημερινή συζήτηση. Και σε αυτό κολλάει και η πρόταση του εισηγητή. Γιατί οτιδήποτε θα αλλάξει την κατάσταση στην Φραγκφούρτη, του ζητάνε να το βγάλει. Πρόεδρε, μετά από την εμπειρία μου την πολυετή στα αεροδρόμια, είναι ότι υπάρχει αύξηση της ποιότητας με τον αριθμό των παρόχων. Και αυτό έχει να κάνει και με την τιμή. Και αυτό σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα για τα αεροδρόμια, καλύτερα αποτελέσματα για τους επιβάτες, γιατί είναι πιο καλή ποιότητα και πιο χαμηλό το κόστος. Γιατί ξέρουμε ότι αν δεν είναι καλές υπηρεσίες που παρέχονται, θα τερματιστεί το συμβόλαιο. Πρόεδρε, εγώ το δέχομαι το, τη συμβαστική Α. Μου προκαλεί κάποια προβλήματα, δεν λέω, αλλά οι υπόλοιπες συμβαστικές μου φαίνονται πάρα πολύ ασαφείς για, την, ε, για τον τερματισμό της μονοπωλιακής θέσης ε, που επικρατεί σε πολλά μέρη στην Ευρώπη. Αν δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του αερολιμένα και των διαφόρων εταιριών και αυτό συμβαίνει μόνο αν, μπουν, αν βγει η λέξη independent από τη συμβαστική α, θα είναι πολύ ασαφές το αποτέλεσμα και κανείς δεν θα τηρήσει τελικά τίποτα. Και στη συμβιβαστική age. Κοιτάξτε, θέλουμε να ορίσουμε εμείς από τον ξελεφάντινο πύργο της Ευρώπης πώς θα ισχύσουν οι λεπτομέρειες σε κάθε αερολιμένα. Νομίζω ότι ούτε την τεχνογνωσία έχουμε, ούτε νόημα έχει. Για τη συμβαστική Α, λοιπόν, Πρόεδρε, την υποστηρίζω, αλλά για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να συγκεντρώσω την υποστήριξη της ομάδας μου. Ευχαριστώ, κυρία Βίλης. Σα ευχαριστώ. 3.000 απασχολούμενοι του προσωπικού εδάφου από πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατήλωσαν σήμερα στην πλατεία Λουξεμβούργου σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Το ανέφερε και ο κύριος Μαν. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην υποστηρίξετε την πρόταση κανονισμού της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να επαναπευθεί. Γιατί χρειαζόμαστε ε, κοινωνικές υπηρεσίες ε, εδάφους και αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οδηγήσει σε, σε χειρότερα εργασιακά σε χειρότερε εργασιακέ συνθήκε και μείωση τη ποιότητα. Οι συμβιβαστικέ προτάσει επιδεινώνουν ακόμα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών με μετακπαίδευση, κατάρτιση των εργαζομένων και δεν θα πρέπει να υπάρχει dumping σε ό,τι αφορά του μισθού. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Ένα κριτήριο για την ανάθεση θα πρέπει να είναι και οι συλλογικέ. Ε, συμβάσεις εργασίας σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των υπηρεσιών σε άλλη υπηρεσία παροχής τέτοιων υπηρεσιών θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τη νομική διάκριση ε, δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε ό,τι αφορά τις εταιρείε υπηρεσιών εδάφους. Δεν ε, περιέχονται προδιαγραφές προστασία κοινωνικής και γι' αυτό λοιπόν ψηφίζουμε, θα ψηφίσουμε κατά. Ο κύριο Γκρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα χαιρόμουν ε, για τις ε, διάφορες ε, συμβαστικές τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση μετά από την αυριανή ψηφοφορία. Θα ήθελα μόνο τρία σημεία να εξετάσω. Καταρχάς, το γεγονός ότι όταν συζητάμε την απελευθέρωση της αγοράς όπως το θέμα αυτό, νομίζω ότι ένα πράγμα ξεχνάμε, ότι ανοίγοντα την αγορά, το θέμα δεν θα πρέπει να είναι η μείωση της ποιότητας και των μισθών, αλλά ότι με το άνοιγμα των αγορών θα πρέπει να πετύχουμε και το αντίθετο. Εγώ είμαι από μια χώρα όπου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ισχύουν και η ποιότητα και η ενίσχυση της ποιότητας, αλλά και η ελάχιστη μισθή. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια εγγύηση για την μη επιδείνωση των μισθών, γιατί όταν υπάρχει μονοπόλιο ή μια παρόμοια κατάσταση σε μια χώρα που δεν υπάρχουν κοινωνικά δικαιώματα και ελάχιστη μισθή, ουσιαστικά δεν, περιορι... δεν ε, βελτιώνεται οι εργασιακές συνθήκες των εργαζόμενων. Το δεύτερο που ήθελα να πω. Νομίζω ότι χθε μιλήσαμε για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αύριο θα μιλήσουμε για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στο συνδρομικό κλάδο και ουσιαστικά θα ακούσουμε διάφορες απόψεις από διάφορες περιφέρειες. Ε. Και αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νομίζω ότι ο συνάδελφος Σεσάρα που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και έδειξε διάθεση σε βασμού Η αλήθεια είναι μεταξύ αυτού και της άλλης ακραίας θέσης. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι το εξής. Δεν είναι δυνατόν αύριο η περιφερειά μου να ψηφίσει απελευθέρωση της αγοράς και σε άλλους ε, τομείς να θέλουμε να προστατεύσουμε τις τοπικές αγορές, για παράδειγμα για το Παρίσι. Δεν μπορεί ο καθένας δηλαδή να ακολουθεί το συμφέρον του. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη του αύριο. Δεν υπάρχει αυτή η λογική λοιπόν στη σημερινή συζήτηση με όλο το σεβασμό προς όλους τους συναδέλφους που προέρχονται από διάφορες ε, περιφέρειες ε, να πω το εξή και για το Hessen και για την Φραγκφούρτη. Με βελτίωση των υπηρεσιών και με αύξηση ενός ευρώ ανά εισιτήριο μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς κατά 5% όλων των εργαζομένων στους αερολιμένες της Φραγκφούρτης. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το πούμε σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτή είναι η Ευρώπη του αύριο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε απλοϊκά επιχειρήματα, τα οποία πολύ απλά δεν στέκουν. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπρόεδρε Βαντάλεν, κάπως παρασυρθήκατε, νομίζω. Έχω 7 αγορητέ στον κατάλογο. Θα αναφέρω τα ονόματα. Και όποιο άλλο θέλει μπορεί να μου πει τι θέλει να μιλήσει. Για να κλείσει τον κατάλογο. Okay. Well, I start with Mr. Liberatsky. Liberatsky πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε, αλλά ίσως να είμαι κάποια από τα αίτια, μία από τις αιτίες της παρεξήγησης. Ας ξεκινήσω όμως με το πρώτο θέμα, αγορά. Αναφέρθηκε κάνα δύο φορές η αγορά. Εδώ δεν μιλάμε για την ευρωπαϊκή αγορά για τις υπηρεσίες εδάφους, μιλάμε για τα αεροδρόμια. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τρεις, θέσεις και παραπάνω πάροχοι υπηρεσιών εδάφου σε ένα αεροδρόμιο και να μπορεί να είναι μια υπερεθνική εταιρεία που να λειτουργεί σε κάθε ε, αεροδρόμιο. Δεν θέλουμε συγκεντρώσεις, αλλά αυτά δεν αναφέρονται στο έγγραφο. Η αύξηση των μισθών κατά 5% στα αεροδρόμια. Πώς ξέρει η διοίκηση των ε, αεροδρομίων. Δεν, δεν προσλαμβάνονται ότι από το ίδιο το αεροδρόμιο αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται. Έχω την εντύπωση ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έπιασε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή τι εννοούμε όταν μιλάμε για υπηρεσίες εδάφους, τι ακριβώς εννοούμε. κατανοώ τα όσα προσπάθησε να πετύχει ο κ. Σάντο, ο Στην Ιαπωνία έχουμε 10 εταιρείε παροχή υπηρεσιών εδάφου στην... στα αεροδρόμια. Σταματά κανεί αυτέ τι εταιρείε από το να μπουν στη Φραγκφούρτη. Μην λέτε ότι υπάρχει μονοπόλιο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτη, διότι ξέρω πώς λειτουργεί. Και ξέρω πώ λειτουργούν και τα μονοπόλια. Πρέπει να παραδεχθώ ότι έχω ανησυχίες όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης. Αντιμετωπίζει εντελώ διαφορετικά τους εργαζόμενους στον τομέα υπηρεσιών εδάφους από τους άλλους τομείς. Αν είχε γίνει σωστή η παρουσίαση, και το κατανοώ σωστά, τότε αυτοί αντιμετωπίζονται εντελώ διαφορετικά. Και πώς θα πετύχουμε τον καθορισμό ελάχιστων αμοιβών. Συμφωνώ με τα υποθέντα του κύριο Βαντάλεν. Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από την πραγματικότητα. Να προσπαθούμε να πετύχουμε φιλελευθεροποίηση και τελικά να καταλήξουμε στα δύο αποτελέσματα όπως και με το πακέτο για τους σιδηροδρόμους. Μην το παίρνετε προσωπικά, κύριε Σιγητά, αυτό που λέω. Αναφερθήκαν κάποια πράγματα. Θέλουμε να επανεξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την πρότασή του. Θα πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ περίεργο ότι κάνουμε μια συζήτηση με ιστορίες που έχει ζήσει ο καθένας σε αεροδρόμια για αποσκευές που χάθηκαν κτλ. Ε, όπως είπε και ο κύριος Γκρός, ε, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να είναι καλύτερη και να μην βασίζεται σε προσωπικές ε, και ιδεολογικές απόψεις. Να συμφωνήσω με τον κύριο Φαντάλενο, γιατί η απελευθέρωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταλήξουμε σε καλύτερη ε, παροχή υπηρεσιών και δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι αυτό ε, ισχύει, γιατί η αγορά αυτή να διαφέρει από όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς κλάδους στην Ευρώπη. Έκανα μια σχετική τροπολογία και βλέπω ότι αποτυπώνεται σε μια συμβαστική πρόταση. Καταλαβαίνω και συμφωνώ για τους τέσσερις αερομεταφορείς αν, ανά μεγάλους αερολιμένες, γιατί θεωρώ ότι είναι βασικό να ανοίξει η αγορά τώρα. Για το θέμα για τα κοινωνικά ζητήματα και τους μισθούς και την ε, εξαγορά ανάληψη ε, προσωπικού. Το αποτέλεσμα θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Δεν με ενοχλεί να οριστούν με τον τρόπο τα κοινωνικά δικαιώματα και με το να απονεμηθεί στους εργαζόμενους αυτά που τους αρμόζουν. Αλλά όταν μιλάμε για κοινωνικά προνόμια, τι να σας πω, αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό, γιατί δεν χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης αυτός ο κλάδος σε σχέση με τους άλλους κλάδους και σε ό,τι αφορά την νομική διάκριση μεταξύ των παρόχων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο και βλέπουμε και στους συνδρόδρομους ότι αν υπάρχει ασάφεια, υπάρχουν βασικά προβλήματα και δεν ε, επιτυγχάνεται η απελευθέρωση της αγοράς και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει νομική διάκριση. Είναι μοναδική εφαρμόσιμη λύση. Νομίζω ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε αυτό το θέμα είναι να κατακαιρματιστεί και τελικά να μην επιτευχθεί η υπεραιτέρω απελευθέρωση σε ό,τι αφορά ε, επίσης, παράλληλα, να εγκριθεί το, 12, το άρθρο 12 της Κοινωνικής ε, Επιτροπής ε, Απασχόλησης, γιατί στην περίπτωση αυτή θα απέχουμε πάρα πολύ από βελτίωση των όρων. Και τελικά θα δώσουμε τροφή σε όσους λένε ότι, κοιτάξτε, δεν λειτουργήσε η απελευθέρωση της αγοράς. Και δεν θα πρέπει να την προάγουμε όπως είπε ο κύριος Γκρός, θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε καλές λύσεις οι οποίες θα είναι εφαρμόσιμες και στην πράξη και σε ό,τι αφορά την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Κράμερ. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν έκανε ανάλυση σφαλμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν αυτό το 80%, 70-80% των επιβατών χάσουν, χάνουν τι αποσκευέ τους και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τις υπηρεσίες εδάφου. Θα ήθελα να ξέρω σε ποιον συμβαίνει αυτό. Εγώ 8 χρόνια ταξιδεύω στις Βρυξέλλε. πότε δεν έχω χάσει τη βαλίτσα. Αλλά οι Άγγλοι μου λένε ότι είμαι αφελής. Στο Χήθρο έχουν 16 οργανώσεις, εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε δύο τέτοιες οργανώσεις. Εγώ δύο παραδείγματα μόνο σας ανέφερα. Μπορούμε να βρούμε και θετικά και αρνητικά παραδείγματα. Θέλω λοιπόν μία ανάλυση. Πού είναι αυτή η ανάλυση. Αν υπάρχουν λοιπόν πολλοί παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για το θέμα αυτό. Θα δημιουργηθεί, χωρίς μία ανάλυση μάλλον, θα επικρατήσει χάος. Δεύτερο θέμα. Ανταγωνισμός είπε ο κύριος Γκρός. Φυσικά με ενοχλεί το γεγονό ότι δεν υπάρχουν ελάχιστοι μισθοί στην ε, Γερμανία, αλλά να θεωρήσουμε ότι μέσω των υπηρεσιών εδάφους θα καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε ελάχιστους μισθούς είναι αφελές. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και θα πρέπει συνειδητά να κάνουμε τα βήματα αυτά. Και αυτό που με απασχολεί και με ε, εκνευρίζει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί αρχές και τελικά δεν επιδρά, δεν επεμβαίνει σε σημείο που θα πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμό. Για το RATP, για παράδειγμα. Roaring Stock στην Γαλλία. σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, απονομή του σχετικού φόρου. Ως ε, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τραστροποιηθεί καθόλου. Και τρίτο σημείο η Ryanair. Στην τελευταία έκθεση επιχειρηματική ε, η Ryanair παρουσιάζει κέρδη 3 εκατομμύρια. Αντικειμενικά έχουν χάσει 5 εκατομμύρια, αλλά επειδή έχουν λάβει 8 εκατομμύρια επιδότηση από εμάς φορολογούμενους, παρουσιάζουν κέρδη. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο και αν τα αντιμετώπιζε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν επίλυε τα προβλήματα αυτά, θα είχαμε βελτιώσει την ε, κατάσταση. Θέλουμε πρώτα απ' όλα ποιότητα και σε θέματα κατάρτισης και σε θέματα εκπαίδευσης και μετά μπορούμε να θέσουμε άλλα θέματα. thank you, Chairman. Κυρία Φώστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Heroic efforts of the are to be... προσπάθειες του εισηγητού είναι πρόσδεκτες. Είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Και πρέπει να επανέλθουμε στο εξή. Έχουμε πακέτο αεροδρομίων. Τρεις εκθέσεις και αυτήν επίσης. Και κατέληξε στα μαύρα της τα χάλια. Ίσως υπάρχουν καλές προθέσεις για βελτιώσεις και το αποτέλεσμα το αντίθετο. Αυτό που θεωρώ απίστευτο είναι το εξής. Σε αυτή την επιτροπή υποστήριξαμε την φιλελευθεροποίηση των αερομεταφορικών εταιριών για πάνω από μία δεκαετία. Στόχος ήταν να απαλλαγούμε από τις κυβερνήσεις να δικούν ε, τις αεροπορικές εταιρείες και να μπαίνουν να αφήνουν εκτός εμπορικές εταιρείες, διότι οι εμπορικές εταιρείες θα πρέπει να δικούν τη βιομηχανία και τις αεροπορικές εταιρείε. Ε, πολλά αεροδρόμια λειτουργούν υπό τον έλεγχο εταιριών και κάποια αεροδρόμια ελέγχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως, συζητούμε κατά πόσο οι υπηρεσίε εδάφου που εργάζονται σε ένα αεροδρόμιο αντιμετωπιστούν διαφορετικά οποιοδήποτε άλλον που εργάζεται σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Αυτό είναι εντελώ παράλογο. Σαν πρώην συνδικαλίστρια που εργαζόμουν στον τομέα των εμπορικών εταιριών, πολέμησα για τι καλύτερε συνθήκε και την καλύτερη αμοιβή για εκείνου ε, με του οποίου δούλευα. Και όταν το κάνει αυτό, αν πάει πληρώσει όσο πιο καλά γίνεται, ελπίζει να έχει καλού εργαζομένου, πιστού και το ίδιο ισχύει και για την παροχή υπηρεσιών εδάφου. Ερώτηση. Πόσοι θα έπρεπε να είναι, αυτό είναι το ζουμί. Ποιο είναι το μήκος ενός ε, σπάγκου. Ε, δούλευα σε ένα αεροδρόμιο που φιλελευθερωποιήθηκε, όπως το Σίπολ που ανέφερε ο Πίτερ, και άλλα αεροδρόμια που έχουν ε, πολλές εταιρείε για υπηρεσίε εδάφους και από παλιά. Υπάρχει και η υπηρεσία αυτοεξυπηρέτηση σε κάποια μικρά αεροδρόμια. Πού φτάσαμε είναι η φρικτή διαφωνία τώρα με την Επιτροπή Απασχόληση που θέλει διαφορετικού κανόνε για εκείνου που εργάζονται σε ένα αεροδρόμιο. Και αυτό είναι παράλογο και γελίο. Τι να πω. Είναι μέλη συνδικάτων. Υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει. Στη χώρα μου απελευθερώσαμε τον τομέα εδώ και χρόνια και έχουμε πολλέ ρυθμίσει εδώ, αυτό με ανησυχεί, που επιβάλλεται σε αεροδρόμια και τα αποτελέσματα είναι αρνητικά όσον αφορά τη λειτουργία του. Στο κάτω-κάτω θέλω να δούμε τι είναι καλό για τους καταναλωτές. Γιατί όλοι φοβούνται τον ανταγωνισμό. Υπάρχει ανταγωνισμός. Λοιπόν, θα έλεγα ότι ο συγητής κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες. Όμως δεν μπορούμε να συζητάμε τον κανονισμό. Ζητώ συγγνώμη του Γερμανού ε, συναδέλφου. Η συζήτηση μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το αεροδρόμιο τη Φραγκφούρτη. Ξέρω ότι είναι θέμα. Ε, το κατανοώ σε, δεν μπορούμε σε επιτροπή να συζητούμε και όλα να στρέφονται γύρω από ένα αεροδρόμιο μιας χώρας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να βρούμε κάποια ρύθμιση. Το καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά δεν κρίνω κι εγώ, δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος για τη Φραγκούρτη. Αύριο στην ψηφοφορία, τι θα γίνει. Όπω υπόθηκε, θα την υποστηρίξουμε την έκθεση. Χρειαζόταν ενδελεχέστερη ανάλυση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν προβάλλει πρόταση ε, σε αυτή την επιτροπή μαζί με τι άλλε εκθέσει. σω περί αυτού πρόκειται. Δεν βλέπω. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Τι βελτίωση έχουμε επιφέρει και το κουβεντιάζουμε έξι μήνε. Καταστροφικά αποτελέσματα. Αποκλίνουσε απόψει. Περί Δηλαδή Δηλαδή εταιρείε να είναι τρει αντί για δύο. Θέλουμε ο καταναλωτή να ωφελείται. Να είναι πιστό στι αεροπορικέ εταιρείε και στα αεροδρόμια καταναλωτή. Λοιπόν, ή θα είμαστε ανοιχτοί και θέλουμε να δουλεύουμε σωστά ή δεν είμαστε τίποτα. Επόμενο. Ο κ. Ντεμπάκ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω, μιας και δεν είμαι από τη Γερμανία και δεν με απασχολεί τόσο πολύ η Φραγκφούρτη, όχι πιο πολύ από κάθε άλλο αεροδρόμιο. Ε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας δυσκολεύει όλους και ο συγητής το δεν ε, δυσκολεύτηκε και αυτός αρκετά. Καταλαβαίνω και αναγνωρίζετε τον κόπο του. Οι συνάδελφοι Μαν και Κλίνσε μίλησαν για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αεροδρομίων. Θεωρώ ότι δεν ήταν ισορροπημένη η πρόταση η οποία έγινε και δεν είμαι ο μόνος που διστάζω σε ό,τι αφορά μια τέτοια ευρία απελευθέρωση σε πολλές συζητήσεις όπως ο Ματιού Γκρός ε, διαπιστώνω ότι σε τομείς όπως ο σιδηρόδρομος, όπως τα ταχυδρομεία, πάντα ταλανίζονται την τομείς αυτή από τα ίδια προβλήματα και νομίζω ότι πρώτα θα πρέπει να κοιτάξουμε το κοινωνικό πλαίσιο πρωτού μιλήσουμε για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς. Αντιθέτως, περαιτέρω α, άνοιγμα των αγορών οδηγεί σε dumping και σε καταπίεση των δικαιωμάτων των απασχολούμενων. Ξέρω ένα αεροδρόμιο σε μία μικρή χώρα που έκλεισε η δεύτερη εταιρεία υπηρεσίες, ε, παροχής υπηρεσιών εδάφους και αναγκαστικά γίνεται διαρκώς διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός αυτός ο σκοπό έχει να κρατήσει υποπίεση την πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά τα πρότυπα. Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σε ό,τι αφορά τα κλινικά πρότυπα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή πρωτοπουλία στον τομέα αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ρίξει τα πρότυπα σε χώρες που επικρατούν υψηλά πρότυπα και να μην βελτιώσει τα πρότυπα σε άλλες χώρες που υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Κύριε Στεγκάλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι σε θέματα απελευθέρωσης τη σχετική συζήτηση δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα λέγοντας ότι αντιμετωπίζουμε τα ίδια θέματα στους σιδηροδρομούς. Ε, δεν είναι το ίδιο. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι μεταξύ Φραγκφούρτης και Αμβούργου, μεταξύ Παρίσι και Άμστερνταμ υπάρχουν πιο πολλά τρένα. Και όταν υπάρχουν πιο πολλά τρένα θα υπάρχουν και πιο πολλοί επιβάτες, γιατί θα είναι καλύτερη η προσφορά. Αλλά αν αυτό είναι ο λόγος ε, να αυξήσουμε τις υπηρεσίε εδάφου και τις σχετικές εταιρείε, τι να σα πω, θα αυξηθούν οι επιβάτες. Δεν υπάρχει σύνδεση, δεν υπάρχει σύγκριση σε ό,τι αφορά την όλη προσέγγιση της απελευθέρωσης, να μην κρίνουμε ανώμια πράγματα. Η συζήτηση ενίσχυσε την πεποίθησή μου ότι καλύτερα να αφήσουμε το νομικό πλαίσιο ως έχει για την κοινωνική πτυχή να πω το εξή μόνο. Οι, υπηρεσίε εδάφου έχουν απελευθερωθεί εδώ και καιρό. Να δείτε τι γίνεται και από πλευρά ε, μισθών. Και σε ό,τι αφορά τη Φραγκφούρτη. Να δείτε τι ποσά καταβάλλονται. Αυτό για όσους θεωρούν ότι πρόκειται να είναι θετικές οι εξελίξεις. Και επειδή έχουν ακουστεί τα υπόλοιπα επιχειρήματα, θα ήθελα να καταλήξω και εγώ στο συμπέρασμα ότι επειδή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αύξηση της ποιότητας με την αύξηση των ε, εταιριών, αυτό είναι το βασικό θέμα. Δεν εγγυόμαστε την αύξηση της ποιότητας με την αύξηση των εταιριών. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα απορρίψω το θέμα αυτό και για το οικονομικό στοιχείο. Το έχω πει και σε άλλες συναντήσεις. Υπάρχουν και μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου σε περίπτωση απελευθέρωσης δεν θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα αναεργαζόμενο θα μειωθεί σε περίπτωση υπερβέρα απελευθέρωσης. Και γι' αυτό λοιπόν ε, σύμφωνα με τον Σνάλφο Μπαχ και θέλω να επαναπεμφθεί η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι παράλογη η κατάσταση. Στις περισσότερες γλώσσες που χρησιμοποιούμε χρησιμοποιούμε τη λέξη αεροδρόμιο, airport, αεροπουέρτο, αερολιμίν, με άλλα λόγια. Και απορρίψαμε μια πρόταση οδηγίας για την φιλελευθεροποίηση των έργων στα λιμάνια, στους λιμένες, διότι θα μπορούσε να διαταράξει τις συνθήκες εργασίας και κατά πολύ. Και δεν ήμασταν σίγουροι ότι η απελευθέρωση των λιμένων θα έδινε προστιθέμενη αξία στους πελάτες. Αυτό κάναμε τότε. Και εγώ είχα μια μικρή εταιρεία, τη χειριζόμουνα, με 100 εργαζόμενους. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ερχόταν μια ομάδα νέων εργαζομένων να εργαστεί και να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό και αν είμαι υποχρεωμένος να τους απασχολήσω θα αντιμετώπιζα πολλά προβλήματα. Αντίθετα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα. Πρέπει να κανονίσουμε κοινωνικά πρότυπα, ποιότητα υπηρεσιών παρέχονται και μετά να βρούμε πώς θα πετύχουμε το στόχο. Όπως είπε και ο προλαλής σας, πρώτα πρέπει να έχουμε πραγματική υποστηθέμενη αξία. Δεν αναφερόμαστε στις χαμένες αποσκευές, μόνο αυτό, αλλά αν έχουμε τέσσερις εταιρείες στη Φραγκφούρτη στο αεροδρόμιο τη Φραγκφούρτη, που είναι τεράστιο αεροδρόμιο. Έχει, έχει διαδρόμους 4,5 χιλιόμετρα. Και αν πάω να παραπονεθώ στον έναν και πω ότι έχασα αποσκευέ και με στείλει στον άλλον, θα πρέπει να φτάσω στην άλλη άκρη. Και δεν θέλω να καταλήξουμε σε κατάσταση όπως έγινε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην κατάσταση στην οποία κατέληξε το Ηνωμένο Βασίλειο με τη φιλελευθερωποίηση που καταμακετίστηκαν οι υπηρεσίε συνδρόμων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν θα ήταν ε, τίμιο. Πιστεύω ότι. Σε σχέση με την απορρίθμιση θα δούμε το κατά πόσο είναι δυνατόν να πετύχουμε αυτού του είδους το συμβιβασμό των θεμητών συμφερόντων των αεροδρομίων ή κατά πόσο θα μπορέσουμε να περιχαρακώσουμε και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Δυστυχώς εδώ πέρα έχουμε κάποια σύγκρουση συμφέροντων και, και τα δύο όλα δεν μπορούμε να τα δεν μπορούμε πετύχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολά και τον ε, σκύλο χορτάτο. Όχι, εγώ δεν θα επικρινώ σε κανένα σημείο τον ε, εισηγητή, όμως έτσι θα γίνει. Και όμως πρέπει να διαλέξουμε Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν είναι δυνατόν να, να, να, να, προχωρήσουμε εάν ό,τι κάνουμε καταλήξει στο να μας καταλήξουν για οπισθοδρόμηση, πισωγύρισμα κλπ. κλπ. Θέλω να την ωφελήσουμε ε, όσο μπορούμε επι, και κλπ. κλπ. Στο πριν λέει το λόγο ο κύριος Μπόλμου, λέω πρώτος, για να δούμε, το ότι σήμερα στη συνάντηση όλοι συμφωνείτε στα εξή δύο. Τόσο νομόφωνοι, σχεδόν ομόφωνα ε, πρεσβεύεται η ευρεία πλειοψηφία πρώτα-πρώτα το ότι τα πράγματα επιδέχονται έχονται βελτίωση με τις πλήρες εδάφου και δεύτερον ότι το αεροδρόμιο του Χήθρο δεν είναι το αγαπημένο σας αεροδρόμιο. Κύριε Μπόλγκουν. To comment on either of your Thanks Σας ευχαριστώ, λέει η Επιτροπή. Άκουσα μεγάλη προσοχή την ε, Επιτροπή σας και από ό,τι βλέπω ε, έχουμε μάλλον στενά περιθώρια στο να τα βρούμε και εμείς θεωρούμε ότι η συμφωνία ε, θα πρέπει τελικά να, να, να, έχει σαν χαρακτηριστικό την ισορροπία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τη βρούμε αυτή την επιθυμητή ισορροπία και ευχαριστώ όλους από όλες τις επιτροπές, εσάς, της ιστορικής αγοράς, απασχόλησης, όλοι οι οποίοι καταβάλλατε τόσο προσπάθειες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο ισορροπία. Έχω κάποιες ε, σύντομες ε, ε, παρατηρήσεις, πρώτα απ' όλα να σας πω και ξανά το εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον αφορά τις υπηρεσίες εδάφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπω ξέρετε θέλουμε με μεγάλη προσοχή να προχωρήσουμε σε κάποιο είδους ε, αύξηση των περιθωρίων επιλογής, ε, να έχουν δηλαδή στο μεγάλο αεροδρόμιο πάνω από δύο, να έχουν τρει υπηρεσίε και επίση να έχουμε και κάποιε διατάξει για τους εργαζόμενου. Ε, και οπότε θα πρέπει να εξορροπήσουμε το ένα θέμα που συνέβρα με το δεύτερο. Πάρα πολύ σωστέ οι τροπολογίε που λέτε στο παράρτημα, δηλαδή για τα ελάχιστα ποιοτικά περιθώρια και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να καθοριστούν σε περιθώριο, σε συγγνώμη, σε επίπεδο ευρωπαϊκό και να δούμε πώ δεν θα έχουμε τελικά κατάδημη τη αγορά υπηρεσιών εδάφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πώ θα έχουμε δίκιο στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών που θα ασχολούνται με τι υπηρεσίε εδάφου και εν τέλει ευχαριστούμε ε, του ε, όσους ανέφεραν για τα κοινωνική επιτυχία, γιατί και εμεί πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πολλά να κερδίσουν από αυτή την αναπλήρωση να, να σας πω ορισμένες μόνο από αυτές τις ε, έχουμε τις αρχές οδηγίες για πρώτη φορά, έχουμε για την ε, μετάθεση, για την κατάρτιση των εργαζομένων με κάποιες διατάξεις και επίσης την υποχρέωση των κρατών μελών του, των κρατών μελών να ελέγχουν τις εταιρείε για τις δεξιότητες, την εμπειρία, ε, τα, προσόντα των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείε και ευχαριστούμε που θα συνεχίσετε μαζί μα για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ανταγωνιστικά αεροδρόμια στην Ένωση και πιο ανταγωνιστικά ιδίω όσον αφορά τι υπηρεσίε εδάφου. Οπότε, με δύο λόγια να δούμε. Ε, αυτές πολλά έχετε πετύχει, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ε, συμφωνήσατε για το άνοιγμα τη αγορά στα μεγαλύτερα αεροδρόμια και επίση ε, δώσατε ευελιξία στα κρατημέλη του να επιβάλλουν κάποια μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα και ιδίω όσον αφορά την μετάθεση των εργαζομένων. για αυτή την μετάθεση απόσπαση μετακίνηση εργαζομένων θα πρέπει να δούμε το πώς θα βελτιωθεί ο σχετικό συνδεσμός για να υπάρχει, υπάρχει επιθυμητή ισορροπία στη συμβαστική ρύθμιση. Ο εισηγητή, σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν θέλω να κολλήσουμε στο ίδιο και στα ίδια σημεία, αλλά θα πρέπει να σας πω έτσι εν συνόψη μια σύνδεση σας ακούσαμε. Δηλαδή, διάφοροι συναδέλφοι το ανέφεραν. Όμως, δεν ξέρω αν είναι όλοι ενημερωμένοι. Δηλαδή, το θέμα αυτό των ελαχίστων προδιαγραφών ποιότητα, θέμα για το οποίο μα μίλησε ο κ. Φαντάλεν, είναι κάτι το οποίο δεν θα το ορίσουμε εμείς. Θα γίνει από το κάθε αεροδρόμιο χωριστά. Όχι, όχι, εμεί εδώ στον Ευβαίνινο πύργο των Βρυξελών δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό. Ούτε εμεί, ούτε η Κομισιόν. Τα αεροδρόμια θα το κανονίσουν αυτό, γιατί τα αεροδρόμια γνωρίζουν τι γίνεται, πόση ώρα απαιτείται για κάθε βαλίτσα, πόση ώρα απαιτείται για κάθε ενέργεια, τέλο πάντων υπηρεσία εδάφου. Κύριε Κράμερ, σα συγχαίρω. Μπράβο σα, σα τυχαίω ποτέ δεν χάσατε βαλίτσα όμω. Στο Βερολίνο το πρωί είχαμε πρόβλημα. Και στο check και αλλού. Δηλαδή, ε, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο ε, υπηρεσιών, εδάφους και άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να χτενίσουμε το έγγραφο και θα μπορέσουμε να τελειοποιήσουμε τους συμβασμούς γιατί η συζήτηση κατέδειξε ότι οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι ε, θεωρούν ότι η απελευθέρωση δεν είναι και τόσο θετική εξέλιξη. Οι σοσιαλιστές επίσης, με τους ελευθέρους και πάλι, ε, επανήλθαν. Ανήκουσαν πρίμνα και είπαν ότι η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική πρόνοια των εργαζομένων δεν προστατεύονται καλύτερα από, ε, από τα όσα λέμε στον έγγραφο. Τέλος πάντων, ελπίζω να τα πάμε καλά. Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε στις 3 η ώρα αύριο και θα ψηφίσουμε και τα άλλα μέτρα, τις χρονοθυρίδες, τα σλότ, το θόρυβο. Και να το που επομένως τώρα περνάμε στην έκθεση Λάκφριντ για τον θόρυβο. Κύριε Αλχαντράουι, σε ποια γλώσσα μας τα πείτε. Αυστριακά, φλαμανδικά, όχι στα αγγλικά, στα αγγλικά λέει, γιατί αντικαθιστά το λέω Λάιχφριντ, κύριε Αλκαντράου. Όπως είπατε, ο κ. Λάιχφριντ δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα εδώ και Ελπίζω να είναι τα θέματα αυτά λιγότερο επίμαχα, λιγότερο να μας διχάσουν από τα θέματα των υπηρεσιών εδάφους. Και την άλλη μεριά ε, θα κολλήσουμε ίσως σε ένα μικρό θεματάκι και θα το συζητήσουμε αργότερα, διότι Έχουμε καμιά 320 τροπολογίες συνολικά, 8 συμβαστικές ο ηγητής και επίσης έχουμε και συμβαστικές τροπολογίες για το γεώμα της έρευνας ελέγχου ε, επίπεδου του, του θορύβου, ενημέρωση, το, το, το πώς θα, θα υπακούν τα αεροπλάνα, γιατί στην αρχική πρόταση της Επιτροπής είχαμε κάποια κενά, γιατί ακριβώς είπαμε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε τι θα γίνουν τα θέματα υγείας και θα πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε την ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων των πολιτών και από την άλλη μεριά του να έχουμε ασφαλεία δικαίου. Όλοι μαζί με την έκθεση, συνεργαστήκαμε θετικά και ο κ. Λάξης περιμένει πώς και πώς να γίνει αύριο η ψηφορία και να είναι αίσιο το αποτέλεσμα και ευχαριστώ τους αδέρφους για την, την, το δομαδικό πνεύμα. Τη συνεργασία. Αυτά είδατε, εγώ σα τα είπα πολύ πιο σύντομα από ότι ο κύριος Σαλάντα. Ο, παρ' όλα αυτά τον ευχαριστώ και εγώ όλους όσους συνέβαλαν ή σε αυτό το αποτέλεσμα. Και βέβαια είμαι έτοιμο να ακούσω όσου έχουν κάποιες παρατηρήσεις και αν χρειαστεί να τα πούμε. Σα ευχαριστούμε κύριε Καντράβη. Γκάλ, Ελκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Λικαντράουι εξ ονόματος του κυρίου Λάιχτφριτ να επιβεβαιώσω αυτά που είπατε ότι πράγματι ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν ήταν ακαθόδες σε αντίθεση με το προηγούμενο. Και ως εκ τούτου νομίζω ότι υπήρξε ευρεία συνένεση και σε ό,τι αφορά τις συμβιβαστικέ προτάσεις. Από τότε που συμφωνήσαμε επί των συμβιβαστικών, ένα στοιχείο με απασχόληση σε ό,τι αφορά το νομικό συμβούλιο. Για τα νέα μέτρα απάλυνσης, όπου στο σημείο 1-2-β αναφέρεται ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα μέτρα για την μείωση του θορύβου. Εγώ από πολιτικής άποψης κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα συνολικό πλαίσιο έξω, από το οποίο θα ε, επιλεχθούν τα πιο αποτελεσματικά μέσα. Αλλά η νομική υπηρεσία μου είπε ότι αν δεν συμπεριληφθεί το θέμα του κόστους, ουσιαστικά υπάρχει ένας αυτοματισμός, γιατί το πιο αποτελεσματικό ασφαλώς είναι να μην υπάρχουν πτήσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρχει καθόλου θόρυβος. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι θα περιοριστούμε μονόπλευρα σε ένα μέτρο και δεν θα εξεταστούν όλα τα μέτρα. Δεν είμαι υπέρ της μείωσης των πτήσεων. Σε καμία περίπτωση. Αλλά, αν παραμείνει η διατύπωση αυτή, προφανώς από ό,τι φαίνεται δηλαδή, οι συνέπειες θα είναι διαφορετικές από αυτές που είχα κατά νου. Γι' αυτό λοιπόν αν θα μπορούσα να κάνω μια τροπολογία μέχρι αύριο για μια αναδιατύπωση Ίσως, ε, εν πάση περιπτώσει, ε, επαναπενθεί η τροπολογία, αλλά μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Κάτι άλλο, στο παράρτημα 2. Θεωρώ ότι κάτι έχει παραμείνει σε δύο σημεία. Στην συμβιβαστική πρόταση έχει παραμείνει η αναφορά για την υγεία, για το όφυλο στην υγεία, αλλά έχει παραμείνει και στο παράδειγμα 1 και στο παράδειγμα 2. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό σας καλώ να το σκεφτείτε και εσείς κατά πόσον αυτό το health benefit, το όφελος ε, για την υγεία, μήπως καλό θα ήταν να αναφέρεται σε ένα σημείο και όχι και στο σημείο 1 και στο σημείο 2. Σκέφτείτε το συνάδελφοι. Μήπως μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τη συμβιβαστική πρόταση. Αυτές τις δύο πάρτρες είχα να κάνω για τις συμβαστικές προτάσεις. Κατά τα άλλα νομίζω ότι και στα βασικά σημεία τα οποία προκάλεσαν τοπικά αναταραχές και στα οποία καταλήξαμε στις συμβαστικές προτάσεις νομίζω ότι οι συμβαστικέ προτάσει είναι προ όφελο όλων. σω όχι προ όφελο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει προ όλων των παραβρισκόμενων. Κύριε Γκάλερ, λέει ο πρόεδρο, δεν ξέρω αν ε, το είπατε όντως, αλλά είπατε ότι θα κάνετε μία προφορική τροπολογία αύριο. Μα κοιτάξτε, εγώ κάποιες φορές ε, λέω να μιλάω αγγλικά για να αποφεύγω τη διερμηνία. Μία προφορική τροπολογία, είπε ο Πρόεδρος, μάλιστα. Αν υποβάλλετε προφορική τροπολογία, ξέρετε ότι ε, μπορεί να υπάρξουν αντιρρήσει. Αν είναι προφορική, εντάξει. Μπορεί να συγχωνευτούν και κάποιε άλλε που αιωρούνται. Και έτσι μπορεί να μην ασπίσουν κι άλλο τα μαλλιά μου τελικά να ακολουθήσω. Κύριο Ντεμπάκερ, για του φιλελεύθερου, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, κύριο Τρεμόσα δεν μπορούσε να έρθει απόψε. Θέλω να ευχαριστήσει τον εισηγητή και του κοιόδη για την έξοχη δουλειά του και τι συναντήσει που διοργανώθηκαν. Είπε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει το δικαίωμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει τη σωστή εφαρμογή ισορροπημένη προσέγγιση και πιστεύει ότι αποτελέχει έγκαιο για του εμπορευομένου και του πολίτε, αλλά καταλαβαίνει βέβαια ότι είναι και μειονοτική η θέση, θέση τη μειοψηφία. Οι περιορισμοί τη λειτουργία δεν είναι μόνη λύση και μπορεί να εφαρμοστούν. Αν πράγματι έχει εμπιστοθεί, υπάρχει πρόβλημα το θόρυβο. Όσον αφορά τα βασικά θέματα τα οποία ετέθησαν, δηλαδή πώ μετρά το θόρυβο, ψηφοεπιδόσεις στο ρίβου ή με τα, τύπου αεροσκαφών. Και τα μέτρα δεν πρέπει να διαφοροποιούνται, πιστεύει, με τα είδη αεροσκαφών, διότι το είδο αεροσκαφών δεν αντιμετωπίζει τι επιδόσει θορύβου, διότι ποικίλει ο θόρυβο σημαντικά για τον ίδιο τύπο αεροσκάφου για πολλού λόγου. Όπω η ηλικία. Κοιτάξτε, ανάβει από του διερμηνεί ένα φωτάκι. Πάτε πολύ γρήγορα. Προσπαθώ να μιμηθώ τον κύριο Τρεμόζα, λέει χαριτολογώντα ο μιλητή. Ε, λοιπόν, και το εκτιμώ ότι προσπαθείτε να τηρήσετε και το χρόνο, λέει ο πρόεδρο, αλλά εδώ αναβοσβήνει το φωτάκι και μου σπάει τα νεύρα, δεν μπορώ. Είστε τυχερό που δεν μιλάω Ολλανδικά, διότι θα ήμουν ακόμα γρηγορότερο. Εξακολουθεί να χαριτολογεί ο μιλητή. Λοιπόν, όσον αφορά τη συλλογή των στοιχείων, ο κύριο Τρεμόσα είπε ότι θα ακολουθήσει προσεκτικά την όλη διαδικασία, την παρακολουθήσει, δεν θέλει να υπάρχει επικάλυψη και αύξηση γραφειοκρατία διότι οι κατασκευαστές αεροσκαφών ήδη δίνουν τα αναγκαία στοιχεία για ε, την χρήση μοντέλων. Στην, ε, στο μοντέλο θορύβου της FAA και όσον αφορά τη διαδικασία θα ήθελα να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή της διάταξης θα πρέπει να είναι σωστή με αποτελεσματικό τρόπο όσον αφορά το κόστος και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Και η ESA να αναφέρεται στους διεθνείς κανόνες την επαλήθευση των δεδομένων. Τέλος, ο κ. Τρεμόσα λέγει ότι δεν του αρέσει η έννοια της αποδοτικότητας που αναφέρεται, προτιμά την σχέση κόστος-οφέλους, ποιότητα ζωής που αναφερόταν στην έκθεση κόστους-οφέλους και ανησυχεί για την έλλειψη αντικειμενικότητας όσον αφορά τις αναφερόμενες πτυχές, πώς προσμετρώνται διότι σε τοπικό επίπεδο έχουν θεθεί στόχοι όσον αφορά τη μείωση του θορύβου και λέει ότι κάθε αεροδρόμιο πρέπει να θέσει τους στόχους όσον αφορά το θορύβο. Η Άλτε δεν μπορεί λοιπόν την συμβαστική 1 και τη συμβαστική 7 να τις υποστηρίξει, αλλά προσβλέπει σε περαιτέρω αγαστή συνεργασία ε, και προσβλέπει σε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Φώστα, έχει το λόγο. Κυρία Φώστα δείχνει κάποιον άλλον. Α, σας ξέχασα. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή που κατέβαλε προσπάθεια για συμβαστικέ προτάσει. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι η πρόταση, η παράγραφος 10, αποτελεί το ακαθόδε ζήτημα. Γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι σε εθνικό επίπεδο να επιτευχθούν ε, συμβιβασμοί για τέτοιους περιορισμούς. Και επειδή ξέρω πόσο αδύναμη είναι η θέση στο συμβιβασμό αυτό, πόσο δύσκολο είναι και πόσο χρησιμοποιούνται και προσωπικά μέτρα πίεσης, πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι θα ήταν λάθος από ευρωπαϊκής ε, πλευράς να προσπαθήσουμε να επιβληθούμε μόνο επειδή προκύπτει κάποιο οικονομικό μειονέκτημα. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι αποδεκτό. Δεν είμαι μεγάλη υποστηρικτρία τη επικουρικότητα τα πάντα. Θεωρώ ότι σε πολλού τομεί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκού κανόνε. Στον τομέα αυτό θεωρώ ότι διαμορφώνεται και ω εξή η κατάσταση. Είναι πολύ διαφορετική η όρη οι συνθήκες που επικρατούν ανά περιφέρεια σε ό,τι αφορά τα επίπεδα θορύβου, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον κτλ. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δεύτερο σημείο, η balanced approach όπως ονομάζεται, η ισορροπημένη προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η προστασία της υγείας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σεβαστό στην τελική ανάλυση δεν ε, χωράει διαπραγμάτευση, μεγάλο κέρδος, λιγότερη προστασία της υγείας. Όταν μιλάμε για προστασία της υγείας και μιλάμε για θέματα υγείας σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τον θόρυβο τη νύχτα και είναι αποδεδειγμένα όλα αυτά, ε, όταν μιλάμε για θέματα υγείας δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτό με το επιχείρημα κέρδους ενός αρλημένα. Δεν είναι αποδεκτός αυτός ο τρόπος εξέτασης των θεμάτων και τι θα λέγατε αν μια μεγάλη ε, επιχείρηση, για παράδειγμα παραγωγής τροφίμων, μέσω προσθήκης ε, ενός ε, τροφίμου επιτύχανε μεγάλα κέρδη, τα οποία θα με έβλεπαν εμένα ως καταναλωτή. Το δεχόμαστε αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό λοιπόν είναι πολύ προβληματικό. Τέλος, ε, τρίτο σημείο μάλλον. Cost efficiency και health efficiency. Θα πρέπει να πούμε το εξή Όταν μιλάμε για cost efficiency, αν αυτό είναι που μετράει, τι θα γίνει σε ό,τι αφορά τον θόρυβο. Θα προσθέσουμε ένα 20%. Και αυτό μπορεί να ωφελέσει ίσως ε, και κάποιες νότιες ε, χώρες. Τι είναι πιο αποτελεσματικό, να υπάρχει ένα καλό παράθυρο προστασίας και τα υπόλοιπα να μην μιλάμε. Γι' αυτό λοιπόν στο σημείο αυτό θεωρώ ότι δύσκολα μπορούν να αφαιρεθούν όλα αυτά τα στοιχεία μόνο και μόνο για να πετύχουμε την βελτίωση του κόστους. Δεν είναι αυτόματα η μείωση του λειτουργικού κόστους το πιο φτηνό, γιατί φυσικά υπάρχει μια διαδικασία σε ό,τι αφορά τις ώρες λειτουργίες του αεροδρομίου. Υπάρχουν και σχετικές νομοθεσίες. Κοιτάξτε, αυτή την τροπολογία, την προφορική, δεν θα την υποστηρίξω. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το συμβιβασμό αυτό. Και όταν με μια προφορική τροπολογία ερχόμαστε και καταρρύπτουμε την ισορροπία της τροπολογίας και του συμβιβασμού, θεωρώ ότι αυτό είναι προβληματικό. Το βασικό για μένα είναι τα δικαιώματα αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ιδάλλως θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλούς συμβασμού. Ευχαριστώ. Και τώρα, κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Well, I think we started... Νομίζω ότι ξεκινήσαμε σε με επικοδομητικές ε, συναντήσεις με τους κοιόδης εδώ και μερικές μέρες. Και ευχαριστώ τον κύριο Λάικφριντ που απουσιάζει. Κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Με εκπλήσει το ότι όλοι στην Επιτροπή επεκρίναμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την οδηγία που ήθελε να την κάνει κανονισμό, άνευ συζητήσεως μαζί μας. Και φαίνεται ότι είμαι η μόνη εδώ που λέει γιατί υποστηρίζουμε έναν κανονισμό όταν επρόκειτο περί οδηγίας και θα μπορούσε να συνεχίσει τούτο τρόπος. Υπάρχουν θέματα επικουρικότητας όσον αφορά αποφάσεις περιθωρίβου, περιαρολιμένων και λειτουργίας αυτών. Δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να συμμετέχει ζητήσει όσον αφορά τη λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ήταν βασικό θέμα για μας και φαίνεται τελικά να το έφαγε μαύρη τρύπα. Αυτά τα είπα έτσι. Προχωρούμε. Ο κύριο Λάικφριντ πραγματικά προσπάθησε να καταλήξει σε Υπέβαλα αρκετέ τροπολογίες κι εγώ. Κάποιοι συμβιβασμοί είναι καλοί και κάποιοι όχι. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα για μας. Όχι όσον αφορά το βασικό θέμα, αλλά συμβαστική ένα, που αφορά άρθρα και παραρτήματα. Το ότι τα θέματα υγείας. Όταν κάποιο ζει κοντά σε αεροδρόμιο και εγώ είμαι στο πιο πολυάσχολο αεροδρόμιο στον κόσμο, στο Χήθρο. Βέβαια έχει τόρυβο, άμα είσαι εκεί. Και οι τρόποι αντιμετώπιση είναι σχετικοί και χρειάζεται συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να αναφέρεται η υγεία στον κανονισμό, αλλά στι αιτιολογικέ σκέψει. Δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει το τι προσπαθείς να πεις. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου μας ξέφυγε αυτό. Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Για τους άλλους συμβιβασμούς. Θα πρέπει να υπάρχουν λειτουργικοί περιορισμοί. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις και αφορά τη συμβαστική ε λατινικό. E. εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετεί, υιοθετεί κατά εξουσιοδότηση πέρα από τα θέματα για τεχνολογικές προσαρμογές. Το Συμβούλιο μετακινήθηκε αρκετά. Υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο ακολουθείται ρεαλιστική προσέγγιση, διότι θέλουμε να λειτουργεί το σύστημα. Πέραν αυτού θα δούμε τι θα γίνει αύριο στην ψηφοφορία. Και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία δεν εξαρτάται από ότι δεν εργάστηκε άοκνα ο εισηγητή. Είναι Αυστριακό. Τεράστιε ομάδε πιέσει στην Αυστρία. Και ο κακομήρη ο εισηγητή κατακλείστηκε από τι πιέσει. Και εγώ το ίδιο από τα διάφορα λόμπι ε, μου είπε ότι κατακλείστηκα από email. Και εγώ δεν τα έλαβα αυτά. Έχει τεράστιες πίεσεις, δεχτεί και τεράστιες πίεσεις για να περάσει αυτό και να συμβιβαστεί. Έχουμε διεθνείς προδιαγραφές. Ξέρουν οι κατασκευαστές ποιες είναι οι προδιαγραφές, οι αεροπορικές εταιρείες, επίσης υπάρχει ισορροπημένη προσέγγιση, συμμορφώνονται άπαντες. Υποστηρίζουμε και τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, ελπίζω. Μπορούμε να τα λύσουμε τα θέματα αυτά. Αυτό που δεν τονίζουμε εδώ στην έκθεση είναι η ευθύνη των κρατών μελών και η χρήση της χωροταξίας. Διότι αυτό ήταν το ζήτημα στις συζητήσεις. Διότι τούνται όσοι μένουν σε περιοχέ που είναι κοντά στο θόρυβο. Κάποιες συμβαστικέ τροπολογίες είναι καλές, εξαρτάται πώς θα λάβει η χώρα η ψηφοφορία. Εγώ πίστευα ότι δεν χρειαζόταν αυτή η έκθεση. Δεν χρειαζόταν και το πακέτο για τα αεροδρόμια. Διότι το μόνο που πετύχαμε το τελευταίο εξάμεινο είναι να έχει προκαλέσει χάο και πόνο. Και τελικά δεν νομίζω ότι πετυχαίνουμε κάτι καινούριο. Τι να κάνουμε, εδώ είμαστε, θα δούμε τι θα γίνει αύριο και ευχαριστώ ειλικρινά τον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Baldwin εκ νέου, κυρία Φώστερ, μιλήσατε για τα λόμπι, για τις ομάδες πίεσης. Και έτσι μπορώ και εγώ να πω επί ευκαιρία ότι το lobbying όσον αφορά και τα τρία ζητήματα ήταν πολύ έντονο, για να το πω διπλωματικά και κομψά. Ό,τι σημαίνει αυτό από διεθνείς οργανώσεις αεροπορικών εταιριών μέχρι και τους κατοίκους που ζουν κοντά στα αεροδρόμια. Ασκούνται πιέσεις. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα δεν νομίζω ότι υπήρξε μεγαλύτερη... Μάλλον υπήρξε μεγαλύτερη πίεση από ό,τι θυμάμαι εγώ σαν Ευρωβουλευτής. Κύριε Μπόλτουιν. Κύριε Μπόλτουιν, λοιπόν, είσαστε στη δύσκολη θέση σήμερα. Ποτέ δεν είναι δύσκολη η θέση όταν μιλώ στην Επιτροπή σας. Ακόμα και για το θόρυβο και για ε, το θόρυβο στο αεροδρόμιο. Πόσους πόντους παίρνω. Μισό λεπτό. Ε, λοιπόν. Α, να μαζέψουμε τα αποτελέσματα της ναυτίας των μελών. Έπρεπε να φέρω σακούλα, λέει και ο Μπόλτουιν. Λοιπόν, ε, ελπίζω να τελευταία φορά που θα παρίσταμε εδώ για αυτό το θέμα. Ο θόρυβος από την ενέργεια κυκλοφορία δημιουργεί σχεδόν χημική αντίδραση και πολιτικές πιέσεις. Σε τοπικό επίπεδο ασκούνται οι πιέσεις και σε γενικότερο παγκόσμιο επίπεδο και όλοι αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πιέσεων σε τοπικό επίπεδο και σε γενικό επίπεδο. Συμφωνώ ότι πρόκειται περί επικουρικότητας και της ενδεδειγμένης εφαρμογής της εν λόγω επικουρικότητας. Εδώ υπάρχει αρκετή συμφωνία. Κάποιοι ζήτησαν εθνικέ αποφάσει και συμφωνούμε με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να παίρνει τι αποφάσει εδώ. Το επαναλαμβάνω εκ νέου και συνεχώ. Ακούσαμε διαμαρτυρίε ότι πρέπει να σεβαστούμε τι τοπικέ διαδικασίε για διαμεσολάβηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη και πάλι αυτέ τι τοπικέ λύσει να τι δεχθεί. Το σεβασμό των διεθνών απαιτήσεων. Όπω η ισορροπημένη προσέγγιση του ΙΚΑΟ. Συμφωνούμε με αυτό θέλουμε να δούμε ένα κείμενο που να αντικατοπτρίζει τι εν λόγω ιδέε και τονίζει το ρόλο των κρατών μελών, που φέρουν την μοναδική ευθύνη, αποκριστική ευθύνη για δικαιμενικό καθορισμό και λήψη αποφάσεων για το θόρυβο και τα μέτρα μείωση αυτού. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επαναλαμβάνω για πέμπτη φορά, δεν θα πρέπει να είναι τίποτα παραπάνω από μια τυπική, ε, τυπικός έλεγχος ε, ε, της σωστής εφαρμογής των μέτρων. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε ε, τις εθνικές λήψεις αποφάσεων και θα ήμασταν έτοιμοι να ακολουθήσουμε μια ρήτρα grandfathering η οποία καθιστά ότι οι νέοι κανόνες δεν θα επηρεάζουν ε, τις εθνικές αποφάσεις αλλά λαμβάνονται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τώρα για τη συμμόρφωση των αεροσκαφών. Υπευλήθησαν διάφορες τροπολογίες για να αναβολούν τα πιο αυστηρά πρότυπα που προτείνονται. Εάν το κάνουμε αυτό, σταδιακά και προχωρήσουμε σταδιακά, στερούμε την απόφαση από τι εθνικέ αρχέ. Να εφαρμόσουν το καλύτερο μέτρο που είναι αποτελεσματικό όσον αφορά το κόστο για την εφαρμογή περιορισμών κατά αεροδρόμιο. Πρόβλημα δεν είναι ο ορισμό, αυτό καθεαυτό, αλλά πότε θα ισχύσει. Αναφερθήκατε στα λόμπι. Ξέρω ότι διάφορε οργανώσει εμπλεκομένων εργάστηκαν πολύ σκληρά. Τους πίεσαν και διάφορες εταιρείες αεροπορικές η χρήση της ενίας των περιφερειακά προσαρμοσμένων αεροσκαφών, συμμορφούμενων αεροσκαφών, ε, πρέπει να ενταχθεί στην ισορροπία προσέγγιση. Θέλουν τα κράτη-μέλη σταδιακά να εξαλείψουν τα αεροπλάνα που δεν συμμορφώνονται ε, ή εν μέρη συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές περιθωρίβου, αλλά πρέπει να το προσεγγίσουμε σωστά για να μειωθούν τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει ε, να μην, ε, αν εφαρμόσουμε γενικά και αδιακρίτως τα μέτρα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε προβλήματα σε εκεί που συμμορφώνονται. Τώρα οι της συμπράξει, το συζητήσαμε. Χρειάζονται αυτέ οι πράξει, ούτω ώστε κάποιε διατάξει να μπορούν να επικαιροποιούνται υπό το φω τεχνολογικών εξελίξεων και αυτό αντικατοπτρίζεται και στι προδιαγραφέ του ΙΚΑΟ. Τίποτα άλλο. Μπορούμε να σκεφτούμε περαιτέρω ακριβέστερε μεθόδου για να πλαισιωθεί το όλο εγχείρημα για τις κατεξοδότητες συμπράξεις, αλλά πιστεύουμε ότι μας χρειάζεται γρήγορη διαδικασία για αποφάσεις, για να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές όσον αφορά τις εκπομπές και το θόρυβο. Δύο άλλα θέματα τέθησαν. Πρώτα απ' όλα υγεία και δεύτερον πληροφορίες για το θόρυβο. Ο κ. Λάιφε σωστά τα λέει, πολιτικός πώς. Αυτό το θέμα της υγείας πρέπει να τεθεί. Επιτάπητος συμφωνούμε με τους στόχους του. Το θέμα είναι πώς, πότε τα θέματα της υγείας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερα να προσπαθήσουμε να τα εξετάσουμε κατά τη διάρκεια τη διαδικασία χρηματολόγηση του θορύβου που αναφέρει στην οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Όπω θεσπίζεται εδώ, αν συμπεριλάβουμε εδώ την υγεία σε αυτόν τον κανονισμό, επιχειρησιακά θα υπάρξει αλληλεπικάλυψη, μάλλον, όσον αφορά του στόχου μειώσει του θορύβου στην οδηγία για περιβαλλοντικό θόρυβο. Θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία να διευκρινίσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τη οδηγία για περιβαλλοντικό θορύβο και τη εν λόγω προτάσεω. Τέλο, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη που μια κουβεντούλα τώρα για τι πληροφορίε για το θόρυβο. Οι εθνικέ αρχέ θα πρέπει να λάβουν αποφάσει επί τη βάση των στοιχείων. Τα στοιχεία είναι διάσπαρτα. Σαν χαρτοπόλεμο σε όλη την Ευρώπη. Σε κάθε αεροδρόμιο δίνονται πληροφορίε σε κάθε πτήση. Απ' την άλλη, έχουμε αεροδρόμια που προσπαθούν να χειριστούν τα τεράστιο όγκο στοιχείων που χορηγούνται. Σκοπό των απαιτήσεων κοινοποίησεω του άρθρου 6 ποιο είναι. Εξορθολογισμό των απαιτήσεων περιθωριβού. Βελτίωση ποιότητα των στοιχείων. Και το Eurocontrol είναι σε άριστη θέση να ασκήσει αυτό το καθήκον. Πιστεύουμε ότι είναι ο πιο πραγματιστικό τρόπο να λύσουν τα πράγματα. Επιμένουμε τι προτάσει μα. Δεν κατανοούμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εξορθολογήσει τι απαιτήσει κοινοποίησεως και προσπαθεί Επίση, να δώσει τα καλύτερα δυνατά στοιχεία στι εθνικέ αρχέ θα πρέπει τότε να καλείται να πληρώσει το λογαριασμό για τι πληροφορίε. Αυτό είναι το ερώτημά μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριο Αλκαντράουι, εκ μέρου του κυρίου Λάιτφριντ, θα είμαι συντομότατο και θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου για τη συνεισφορά του για κάποια ίσον σημασία θέματα. Δεν είναι όλοι πολύ ενθουσιώδεις, αλλά ε, το εκλαμβάνω ως υποστήριξη. Οι περισσότεροι υποστηρίζετε τους συμβιβασμούς. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γκάλερ αν θα μπορούσε, μάλλον θα του ζητήσω, αν θα μπορούσε να μην υποβάλει προφορικές τροπολογίες τελευταία στιγμή. Υπάρχει ακόμα χρόνος, θυμίζω, για την Ολομέλεια για να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα. Είναι πρώτη ανάγνωση. Μπορούμε ε, ακόμα να διαπραγματευτούμε ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ εκ νέου για τα πάντα. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του θέματος. Λοιπόν, αύριο στις 3 θα γίνει ψηφοφορία. Πάρτε τις κάρτες ψηφοφοριών. Πέρα συνεδριέσεως μέχρι 9 την πρωί αύριο, όπου ασχοληθούμε με το θέμα μας, τα ευρωπαϊκά δίκτυα, στην ίδια αίθουσα. Μπορεί να τα αφήσει εκεί και αν κάποιο θέλει να έρθει με κλάρκ, ε, αν τα σηκώσει, α έρθει και να τα μαζέψει. <laughs>